από το ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και το ECR έλαβα προτάσεις για διορισμούς ε, σε επιτροπές και αντιπροσωπείες θα εμφανιστούν στα πρακτικά της ε, Συνόδου και οι παρατηρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις εγκρίσεις των πρακτικών.